Okay. I think it's, it's time to start. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Και, ε, ναι, μεν έχουμε έναν τέταρτο καθυστέρηση, αλλά παρόλα αυτά να σας καλωσορίσω στο τελευταίο τμήμα της συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Όπως ξέρετε, σήμερα δεν θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων με τους επιτρόπους Χόγκαν και Βέστεχερ. Διότι δυστυχώς ε, ε, πρέπει να συμμετάσχουν σε μια σημαντική συνεδρίαση της Επιτροπής. Η Γραμματεία ε, αυτή τη στιγμή διερευνά τις δυνατότητες επανακαθορισμού της συζήτησης μαζί τους. Οπότε, θα περάσουμε στα επόμενα θέματα της σημερινής διάταξης. Έχουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη Δυτική Σαχάρα και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η απόφαση στις ε, εμπορικές συμφωνίες ε, με το Μάροκο, στις συμφωνίες ε, ελευθέρω εμπορίου. Όπως θα γνωρίζετε, η απόφαση αυτή προβλέπει ότι οι συμφωνίες σύνδεσης και φιλελευθεροποίησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκ δεν εφαρμόζονται στη Δυτική Σαχάρα. Το δικαστήριο λοιπόν ακύρωσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου. Σήμερα θα έχουμε μία παρουσίαση από την νομική υπηρεσία Έχουμε λοιπόν τον κύριο Μέντολα εδώ. Μεγάλη μας χαρά. Και να καλωσορίσουμε και τον κύριο Πικέτα που θα μας ε, κάνει μια παρουσίαση από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για το θέμα αυτό. Οπότε να σας δώσω το λόγο χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση για να μας παρουσιάσετε την κατάσταση για το θέμα αυτό. Να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ε, τωρινή συγκυρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω πώς διεξήχθη η δίκη και τι επιπτώσεις έχει αυτή η απόφαση του παρελθόντος Δεκεμβρίου. Ποιο είναι το, ποια είναι η προϊστορία. Έχουμε μια συμφωνία σύνδεσης με το Μαρόκο από το 1996 και το 2010 επίσης συνήφθη μια συμφωνία απελευθέρωσης των συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της από τη μία και του βασιλείου του Μαρόκου από την άλλη, η οποία προβλέπει μειωμένους δασμούς ή κατάργηση των δασμών για κάποια αλλιευτικά και γεωργικά προϊόντα. Η συμφωνία αυτή εφαρμόστηκε για τα προϊόντα από τη Δυτική Σαχάρα. Το 2010, το μέτωπο, 12 ε, συγγνώμη, το μέτωπο Φολισάριο υπέβαλε προσφυγή για την κατάργηση της απόφασης του Συμβουλίου που ενέκρινε αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ένωσης και Μαρόκου. Ένα από τα επιχειρήματα τα οποία παρουσίασε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου το Συμβούλιο για να στηρίξει την συμφωνία είναι ότι όταν συνήφθη οι δύο συμβαλόμενοι, Ένωση και Μαρόκο, είχαν την πρόθεση η συμφωνία να καλύψει και τα προϊόντα του γενικού, συγγνώμη, του, της Δυτικής Σαχάρας. Οπότε το Γενικό Δικαστήριο δεν υπάρχει καμία ρήτρα που να εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει μια συμφωνία σε μια αμφισβητούμενη περιοχή όπως είναι η Δυτική Σαχάρα αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας δεν ε, κάνει διακρίσεις σε βάρος του πληθυσμού της Δυτικής Σαχάρας. Επειδή δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το Συμβούλιο είχε ελέγξει εάν όντω θα εφαρμοστεί η κατάσταση, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της στην ε, Δυτική Σαχάρα. Στις αρχές ε, του παρελθόντος έτους το Συμβούλιο έκανε έφεση κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου και ένα ή μάλλον το κύριο επιχείρημα του, του Συμβουλίου ήταν ότι το μέτωπο Πολυσάριο δεν ήταν ε, διάδικος ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τυπικά ενέκρινε την ε, προσφυγή, την έφεση του Συμβουλίου, αλλά με μια επιχειρηματολογία που τελικά στρέφεται κατά του Συμβουλίου, διότι θεωρεί το δικαστήριο ότι για να διαπιστώσουμε εάν και κατά πόσο το Πολυσάριο μπορούσε να είναι ενάγων ε, ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, θα έπρεπε να ελέγξουμε εάν και κατά πόσο η συμφωνία αυτή με το Μαρόκο μπορεί να εφαρμοστεί στη Δυτική Σαχάρα. Και θεωρεί ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να εξετάσει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου σε συμπεριλαμβανομένης της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών και των σχετικών αποτελεσμάτων των συμφωνιών. Και το δικαστήριο τονίζει ότι σε μία συμβουλευτική απόφαση του 1975 το Διεθνές Δικαστήριο θεωρεί ότι ο λαός της Δυτικής Σαχάρας απολαμβάνει πλήρως του, δικαιωμα... του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Και μία άλλη απόφαση, ένα άλλο ψήφισμα των ΗΕ τόνισε ότι οι περιοχές που δεν αυτοδικούνται έχουν ένα χωριστό και ιδιαίτερο καθεστώς. Και η Δυτική Σαχάρα είναι μία από αυτές τις περιοχές. Είναι στο κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών. Από το 1963. Οπότε, το πόρισμα στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο είναι ότι εφόσον η Δυτική Σαχάρα έχει ιδιαίτερο και χωριστό καθεστώς. Η συμφωνία μεταξύ Ένωσης και Μαρόκου δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη Δυτική Σαχάρα. Διότι είναι χωριστή οντότης. Το δικαστήριο λοιπόν λέει ότι λόγω των σχετικών επιπτώσεων των συμφωνιών παρά την εκτίμηση του Γενικού Δικαστηρίου η συμφωνία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη Δυτική Σαχάρα εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο λαός της Δυτικής Σαχάρας έχει συνενέσει σε αυτήν την εφαρμογή. Διότι, από ό,τι βλέπουμε από τα στοιχεία για την περιοχή, δεν έχουν συνενέσει οι κάτοικοι της Δυτικής Σαχάρας. Άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτούς, σε αυτή την περιοχή, αυτή η συμφωνία. Οπότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου και άρα η συμφωνία απελευθέρωσης ναι με ενισχύει αλλά μόνο υπό τους όρους που αναφέρει στην απόφασή του το δικαστήριο. Υπάρχουν άμεσες πρακτικές συνέπειες γιατί εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου άλλες δύο μάλλον καλύτερα, μία ενώπιον του γενικού και μία ενώπιον του ευρωπαϊκού. Δύο υποθέσεις εκκρεμούν. Και επίσης, θα έχουμε και πολιτικές επιπτώσεις. Αν εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία στη Δική Σαχάρα με διαφορετικό τρόπο, μάλλον για να εφαρμοστεί στη Δική Σαχάρα θα πρέπει να εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι εφαρμόζεται στο Μαρόκο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παίρνω το λόγο σήμερα εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας και θα ήθελα να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό, περιγράφοντάς σας ποια είναι και η στάση της Υπηρεσίας Εξαιρετικής Εξωτερικής Δράσης. Δεν είμαι βέβαια νομικός, ακούσαμε ποια είναι η νομική άποψη μόλις, οπότε η αντιμετώπιση δική μου ε, ουσιαστικά θα ασχοληθεί με το ε, προς τα που πρέπει να κινηθούμε τώρα, ε, μια και έχουμε πλέον τη γνωμοδότηση ή μάλλον την απόφαση του δικαστηρίου και είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με αυτήν. Α δούμε καταρχήν ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Μαρόκο. Είναι μια πολύ σημαντική ε, σχέση. Είναι μια ε, διακεκριμένη εταιρική σχέση η οποία προσφέρει ένα πολύ υψηλό βαθμό και αλληλεπίδραση και συνεργασία σε χώρου στρατηγικού για εμάς, όχι μόνο δηλαδή σε οικονομικά θέματα ή σε εμπορικά θέματα, όπου είναι πολύ σημαντική η σχέση που έχουμε τη χώρα αυτή, αλλά παράλληλα και για μια σειρά από άλλε πολιτικέ, οι οποίε είναι προ το αμοιβέ μας συμφέρον, το περιβάλλον, το κλίμα. Ε, ξέρετε πώς η τελευταία κόπ συνεδρίασε στο Μαρακές ε, πέρσι, στα τέλη της χρονιάς. Μας συνδέουν ε, κοινά συμφέροντα στον χώρο της ασφάλειας, της περιφερειακής σταθερότητας και βέβαια Υπάρχει και το πολύ μεγάλο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής. Οπότε είναι μια ευρύτερη σχέση, ε, πολύ βαθιά και θα πρέπει κανείς να είναι ειλικρινής και να πει πως το τελευταίο έτος, ενάμιση έτος, έχουμε υποφέρει σε κάποιο βαθμό από την υπόθεση που συζητάμε σήμερα, αλλά και από άλλες δύο υποθέσεις που αυτή τη στιγμή εκκρεμωδικούν στο δικαστήριο. Πρώτον, του ποια είναι η σχέση της Δυτικής Σαχάρας μέσα στο πλαίσιο της συμβατικής εταιρική σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου είναι μια υπόθεση η οποία έχει επιβραδύνει την εμβάθυνση της ε, εταιρική αυτής σχέσης στο βαθμό που είχαμε πετύχει στο παρελθόν και όπου νομίζω ότι υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία θα πρέπει να επανακάμψουμε. Τώρα η απόφαση του Δεκεμβρίου ήταν απερίφραστη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομική βάση για να εφαρμόσουμε αυτούς τους προτιμησιακούς ε, δασμούς σε προϊόντα τα οποία προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι, να μην υπάρχει καμία παρερμηνία. Αυτό δεν σημαίνει απαγόρευση ε, εισαγωγών προϊόντων από τη Δυτική Σαχάρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, απλώς δεν υπάρχει νομική βάση για να τους δώσουμε αυτούς τους ευρωπαϊκούς προτιμησιακούς δασμούς. Θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση αυτή, να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε, να ξεπεράσουμε το εμπόδιο αυτό μέσα στο όλο πνεύμα της συνεργασίας μας με το Μαρόκο και αυτό που είναι ξεκάθαρο ότι οτιδήποτε θέλουμε να πετύχουμε θα πετύσει πολύ στενή συνεργασία, όχι μόνο σε πολιτικό αλλά και σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ημών. Κάπου βιαζόμαστε. Ε, νομίζω πως βιαζόμαστε περισσότερο λόγω των ε, οικονομικών, ε, της οικονομικής πραγματικότητας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς επιχειρηματίες και εμπορευόμενους που ε, έχουν εμπορικές σχέσεις με το Μαρόκο, με προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα και καταλαβαίνετε ότι για το εμπόριο χρειάζεται σαφές κανονιστικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο και για τους εμπορευόμενους είτε από την μαροκινή πλευρά είτε από την ευρωπαϊκή όλοι χρειάζονται να ξέρουν ποια είναι η δασμολογική πολιτική στην οποία εμπίπτουν ή όχι. Οπότε και στο σημείο αυτό έχουμε και αρκετά ογκώδη αλληλογραφία η οποία μας πιέζει χρονικά ζητώντα μας να διευκρινίσουμε αυτά τα θέματα. Επιθυμούμε να βρούμε μια λύση η οποία θα διατηρήσει τις πρακτικές στις οποίες είχαμε καταλήξει στο παρελθόν και που δεν θα επιβάλλει κάποιες κυρώσεις σε όσους εμπορεύονται με τη Δυτική Σαχάρα. Δεν θέλουμε με τον τρόπο αυτό να βλάψουμε όσους ζουν στην περιοχή αυτή, ούτε τους ε, εμπορευόμενους από τη Δυτική Σαχάρα. Άρα θέλουμε να δημιουργήσουμε μια άλλη νομική βάση που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Βεβαίω θα πρέπει να συμμορφωθούμε με την ε, αιτιολόγηση της απόφασης του δικαστηρίου. Δεν είναι εύκολο, ήταν πάρα πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Και βεβαίω επαναλαμβάνω, υπάρχουν και αυτές οι δύο εκκρεμίε υποθέσεις ακόμα στο ΔΕΚ. Οπότε ό,τι οικοδομήσουμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να προσπαθήσει να προλάβει ε, τα όσα θα εκδώσει για τις επόμενες δύο υποθέσεις του δικαστήριο αργότερα φέτος. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι θα έχουμε μια αυτούσια μεταφορά της πρώτης απόφασης της Οπότε υπάρχει ένας βαθμός αβεβαιότητας, τουλάχιστον νομικής αβεβαιότητας, στις προσπάθειες που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Έχουμε και κάποια άλλα σημεία και αυτό είναι η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο. Θα γνωρίζετε κι εσείς πως αυτή τη στιγμή τρέχει μια ειρηνευτική διαδικασία του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα έτσι ώστε αυτή η σύραξη που χρονίζει να λυθεί με πολύ στεναρή στήριξη αυτής της ε, ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα η πραγματικότητα είναι πως αν ε, δεν την χαρακτηρίσουμε τελματώδη θα μπορούσαμε να πούμε πως την τελευταία δεκαετία οι πρόοδες ήταν εξαιρετικά αργοί. δεν διαφαίνεται κάποια λύση στον ορίζοντα. Παρ' όλα αυτά Στη διμερή απόκριση που θα δώσουμε στη συνέχεια αυτής της απόφασης του δικαστηρίου θα πρέπει να καταφέρουμε τα εξή δύο. Θα ξεκινήσω με μια αρνητική φράση που είναι να μην επιτρέψουμε σε κανένα από τα δύο μέρη ε, ή σε κανένα από τους δύο διαδίκους να βλάψει την ενδεχόμενη κατάληξη αυτής της ειρηνευτικής διαδικασίας και, για να το πω και πιο θετικά, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προτείνουμε μια λύση η οποία θα μπορούσε με τη σειρά της να βοηθήσει ε, αυτή η ειρηνευτική διαδικασία να αναπτερωθεί. Άλλωστε το είπε και ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και έχει πει πως σύντομα θα ξεκινήσει η διαβουλεύση για το θέμα αυτό με τη διεθνή κοινότητα. Λοιπόν, να σας πω, θα πρέπει πως για το θέμα αυτό έχουμε ε, το πλαίσιο του ΟΗΕ, έχουμε το διεθνές δίκαιο με το οποίο πρέπει να συμμορφωθούμε και να τα θεωρήσουμε αυτά ως σημεία εκκίνησης και να σας περιγράψω με πιο συγκεκριμένα βήματα ε, το πώς θα κινηθούμε. Να σας πω καταρχήν πως όπως διαπιστώσατε και εσείς, η συνεργασία μας με το Μαρόκο είναι στενή. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η απόφαση, την 21η Δεκεμβρίου του 2016, ε, εκείνη τη στιγμή ο Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εξέδωσαν μια κοινή δήλωση για το ότι θα εργαστούν για να βρουν την βέλτιστη λύση. Έκτοτε έχουμε προχωρήσει με διπλωματικές επαφές με τους Μαροκινούς που οδήγησε σε μία ε, συνάντηση που έκανε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Μαρόκου με την ύπατη εκπρόσωπο εδώ στις Βρυξέλλες με κάποιες διερευνητικές ε, επαφές για το τι είναι βιώσιμο Βέβαια το σημείο αναφοράς είναι η συμμόρφωση με την απόφαση του ΔΕΚ και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα σημεία κίνησης τα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Αυτό που έχουμε κατά νου είναι να δημιουργήσουμε μία λύση η οποία θα είναι νομικά στέρεη, ε, σφριγιλή, που θα αντιμετωπίσει κάποιες ε, μελλοντικές ενστάσεις ή προσφυγές που δεν θα καταρρεύσει υποπολιτική πίεση σε όλα τα πλαίσια στο οποία θα κινηθεί. Γιατί προσπαθούμε στην συμφωνία αυτή να προχωρήσουμε σε μια ρητή επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης της συμφωνίας έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και τη Δυτική Σαχάρα βέβαια στα πλαίσια μιας νομολογίας η οποία είναι σύμμορφη και ευθυγραμμισμένη με την νομοκλατούρα της, με την ονοματολογία, με συγχωρείτε, των Ηνωμένων Εθνών. Μία ονοματολογία λοιπόν η οποία θα ξεκαθαρίζει στο ότι δεν υπάρχει καμία προκατάληψη προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, ε, ανεξάρτητα με τη νομική ε, λύση που θα επιλέξουμε. Η απόφαση του δικαστηρίου βεβαίως συνοδεύεται από την ε, αιτιολόγηση αυτής και εκεί θα διαβάσατε πως έχει να κάνει με την συγκατάθεση του πληθυσμού της Δυτικής Σαχάρας ένας παράγοντας τον οποίο βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα το κάνουμε με έναν τρόπο ο οποίος σας επαναλαμβάνω νομικά θα είναι ε, στέρεος. Και θα, είναι και, και θα νομιμοποιείται και πολιτικά. Και βέβαια καταλαβαίνω πως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να το συζητήσουμε και να το διαπραγματευτούμε, αλλά επειδή μέχρι στιγμής οι σχέσεις εργασίας που είχαμε σε πρακτικό επίπεδο και στο τεχνικό επίπεδο, όχι μόνο στο πολιτικό, με τις ε, μαροκινές αρχές, μπορώ να σας πω πως είμαι αρκετά σίγουρος πως μπορεί να το οδηγήσουμε σε μια ευτυχή κατάληξη. Έγινε μια πρώτη τεχνική συζήτηση με το Μαρόκο δεν μιλάμε για ε, διαπραγματεύσεις, αλλά για διερευνητικές συζητήσεις. Αύριο θα γίνει μια δεύτερη τεχνική συζήτηση. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε πως αυτές οι διερευνητικές τεχνικές επαφές μας δίνουν μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να εργαστούμε ώστε να καταλήξουμε σε μια πρόταση. Πρόταση την οποία θα υποβάλουμε στο Συμβούλιο έτσι ώστε να μας δοθεί μια εντολή για να διαπραγματευτούμε την νομική προσαρμογή ε, της ε, συνθήκης, της συμφωνίας, ακολουθώντας την συνήθη διαδικασία του άρθρου 2.18 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια θα περάσει και από εσάς το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα να περάσουμε στη συζήτηση. Ο κύριος Μποβέ καταρχάς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Η υπενθύμηση μόνο όταν έγινε η συζήτηση και η επέκταση της Γεωργικής Συμφωνίας ήμουν αρμόδιος εισηγητής από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και ως εισηγητής είχα συστήσει στο Κοινοβούλιο να αρνηθεί τη συμφωνία και να καταψηφίσει στην Ολομέλεια λόγω των νομικών κολλημάτων τα οποία προέκυπταν από την ε, περίπτωση της Δυτικής ε, Σαχάρας. Η νομική υπηρεσία τη θυμάται πολύ καλά αυτή την ε, περίοδο, διότι η συζήτηση διήρκεσε δύο-τρει μήνε και μετά από ενάμιση χρόνο διαφωνούσαν οι διάφορες νομικές υπηρεσίες, το Συμβούλιο από τη μία, το Κοινοβούλιο από την άλλη. Το Κοινοβούλιο ήταν ε, πολύ ε, πιο στέρεο στη θέση του από ότι το Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά όμως αποφασίσατε να ε, προχωρήσετε. Αυτά το οποίο τελικά θα συνέβαινε συνέβη και η απόφαση ακυρώθηκε λόγω μιας περιοχής η οποία αποτελεί μια μη αυτόνομη περιοχή ε, λόγω των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Και τώρα λοιπόν έχουμε περιέχθει σε μια ε, κατάσταση η οποία δεν έχει ξανασυμβεί, μια συμφωνία η οποία δεν μπορεί να προχωρήσει, έχει παγώσει και πραγματικά εγώ ανησυχώ ακούγοντας αυτά που άκουσα σήμερα γιατί δεν βλέπω διέξοδο με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί θέλω να μιλήσουν και άλλοι, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα εσωτερικό ευρωπαϊκό νομικό πρόβλημα. Και αυτό το εσωτερικό πρόβλημα είναι η Ισπανία. Η Ισπανία ποτέ δεν ανέλαβε τις ευθύνες της ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών για την ε, ε, συγκεκριμένη περιοχή, την οποία ουσιαστικά τη θεωρεί απικία της ε, και πρέπει να σταματήσει να, την αποκειοκρατία στη Δυτική Σαχάρα. η η Ισπανία λοιπόν δεν έχει ποτέ κάνει αυτό που τη αναλογεί στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε μια συμφωνία σε μια περιοχή χωρίς αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνο για την απεικιοποίηση δεν να αναλάβει τις ευθύνε του για να ξεκινήσει μια διαδικασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είναι αδύνατο. Και εδώ υπάρχει πραγματικά ε, πρόβλημα δικαίου. Και Υπάρχει το θέμα των Ηνωμένων Εθνών και η ευθύνη της Ισπανίας που πρέπει να ξεκινήσει και τη διαδικασία της απόφασης των κατοίκων της Δυτικής Σαχάρας κατά πόσον θέλουν να είναι εξάρτητοι και επομένως δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Δεν θα αποφασίσω εγώ τη λύση. Οι κάτοικοι θα το αποφασίσουμε και υπάρχουν και ψηφοφορίες κλπ. Και αυτή είναι η διαδικασία. Και γιατί σας το λέω αυτό. Διότι αν δεν γίνει αυτή η δουλειά πώς θα υπάρξει και ε, κάτι σε νομικό επίπεδο για τις εξαγωγές. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση παρά μόνο με ένα εταίρο που είναι το Μαρόκο αυτή τη στιγμή που λέει ότι έχει τη διοικητική διαχείριση της περιοχής αλλά χωρίς κανένα νομικό δικαίωμα και το κάνει απλώς για της βίας. Δεν είναι ε, θέμα κατά της, του Μαρόκου αυτό, αλλά αυτή είναι η νομική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε κάποια προϊόντα τα οποία προέρχονται από την περιοχή, γεωργικά ή αλευτικά, πρέπει να γίνουν τριμερείς συζητήσεις. Και δεν άκουσα τίποτα από εσά ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Άκουσα θα πρέπει κανονικά να έχουμε τους εκπροσώπους της Σαχάρα, εκπροσώπου του Μαρόκου, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις και του Ευρωπαίου εκπροσώπου. Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε διαπραγμάτευση που να μην έχει τα τρία μέρη. Γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό σα είπε, ότι η Σαχάρα δεν είναι τμήμα της Μαροκινής επικράτειας, αλλά λέγοντα το αυτό αναγνωρίζει και την καταγγελία του εκπροσώπου των ε, κατοικών της Δυτικής Σαχάρας, ε, ε, και ε, ουσιαστικά μας καταφέρνει στην αρχή, όπως το καθορίζει και η απόφαση του δικαστηρίου. Πρέπει να κάνετε τριμερείς συζητήσεις και δεν μπορείτε να το παρακάμψετε αυτό. Ε, και το θέμα είναι τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε το μεταξύ. Εγώ το συζητώ, δεν θα γίνει αυτή τη στιγμή, αλλά έχω κάποιες ιδέες επί του θέματος. Πιστεύω όμως ότι καταρχάς θα πρέπει να έχουμε την ειλικρίνεια να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ε, η ε, πρωτίστως ευθύνη της Ισπανίας σε αυτή την περίπτωση. κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης που ήρθαν εδώ να μας διευκρινίσουν λίγο τα πράγματα αυτής της υπόθεσης. Δεν σας κρύβω βεβαίως ότι είναι πολύ περίπλοκο να, να αντιληφθώ ακριβώς την κατάσταση, διότι τελικά το δικαστήριο εξέδωσε μία απόφαση Ε, που φαίνεται να διορθώνει την αρχική απόφαση, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Τελικά λέει ότι δεν εφαρμόζεται στη Δυτική Σαχάρα συμφωνία γιατί δεν είναι μαροκινή επικράτεια. Ε, και δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ε, να σας πω όμως ότι για μένα αυτό που είναι πιο ανησυχητικό ε, από αυτές τις αποφάσεις είναι πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Διότι εδώ υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι είναι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι εμπιστεύτηκαν τη συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και για την οποία γνωμοδότησε και το Κοινοβούλιο και που διεξαγόταν ομαλά, φαίνεται ότι κάλυπτε όλες τις ε, πλευρές, φαίνεται ότι υπήρχε συμφωνία και ξαφνικά βρίσκονται τελικά στο δρόμο. Είναι άνθρωποι τους οποίους πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να ανησυχούμε για αυτούς, είναι γεωργοί, αλληλείς και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση και οι ευθύνε που θα αναλάβουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτούς του ανθρώπου μέχρι να υπάρξει αυτή η νέα συμφωνία. Διότι αν κατάλαβα καλά, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση για μια νέα συμφωνία. Λαμβάνοντας υπόψη και πόσο ε, ε, στοιχίζει να διαπραγματευτούμε ε, νέες συμφωνίες, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα στο οποίο θα υπάρχει νομικό κενό και υπάρχουν οικογένειες εργαζομένων που εξαρτώνται από τη λύση που περιμένουμε να υπάρχει στο συντομότερο δυνατόν. Ε, υπάρχει υποχρέωση για ασφάλεια δικαίου, την οποία αυτοί θεωρούσαν ότι είχαν. Και θα ήθελα να ξέρω λοιπόν το εξή. Ποια είναι η θέση μα, τι θα κάνουμε εμεί στη συνέχεια για να βοηθήσουμε εμεί αυτέ τι ευρωπαϊκέ οικογένειε που ανησυχούν ε, πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ από πλευρά μου θα ήθελα να μου εξηγήσετε δύο πράγματα. Πρώτον, και εδώ θα συμφωνήσω και με τα όσα είπε ο Ζεμποβέ προηγουμένω. Μα είπατε προηγουμένω ότι θα συνεργαστείτε με το Μαρόκο, θα υπάρξει λύση με το Μαρόκο κλπ. Ε, ξεχνάμε όμως ότι υπήρξε και μία απόφαση η οποία αναγνωρίζει δικαιώματα και για τους κατοίκους της Δυτικής Σαχάρας. Δεν θα μιλήσετε λοιπόν με τους ανθρώπους αυτούς για να δούμε πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση. Αυτό είναι το ένα. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω και ε, σε ποιο βαθμό τηρείται η συμφωνία, διότι η απόφαση είναι σαφής. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν εάν κάνετε κάτι για να τηρηθούν τα όσα προβλέπει η συμφωνία ή ε, η απόφαση, συγγνώμη, ή δεν τηρείται τίποτα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί κάναμε την ίδια συζήτηση στην Επιτροπή Αλίας. <clears throat> Κατά τη συζήτηση της Συμφωνίας Σύνδεσης. Η απόφαση έχει επιπτώσεις στις συμφωνίες. να μας εξηγήσουν ποιες είναι ακριβώς αυτές οι επιπτώσεις οι εκπρόσωποι της Κομισιόν και της εξωτερικής δράσης. Δεν είναι οι ίδιες επιπτώσεις στον τομέα της εμπορικής συμφωνίας και στον τομέα της συμφωνίας σύνδεσης. Είναι διαφορετικά τα θέματα. Είναι διαφοροποιημένη η αντιμετώπιση. Το λέω αυτό για να ξέρουμε τι λέμε. Είναι περίπλοκο το θέμα για μένα. Το είπε και η κυρία Εράνθ. Δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είναι οι ίδιες επιπτώσεις. Δεν είναι. Τώρα για τη γεωργική λοιπόν συμφωνία. Από ό,τι κατάλαβα λοιπόν, η γεωργική συμφωνία είναι σαφής. Η απόφαση του δικαστηρίου, κατά τη γνώμη μου, είναι σαφής σε σχέση με τη γεωργική συμφωνία, η οποία λοιπόν ισχύει, αλλά μόνο για την επικράτεια του Μαρόκου, όχι την περιοχή που απλώς δική το Μαρόκο, δηλαδή τη Δυτική Σαχάρα, <clears throat> Δεν είναι όμως ε, η περιοχή αυτή περιοχή του Μαρόκου, αν και τη δική το Μαρόκο. Υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις και με κάθε σεβασμό και αγάπη προς τον κύριο Μποβέ του λέω ότι αυτά που πρέπει να επιλύσει ο ΙΕ να τα λύσει ο ΙΕ. Σας λέω ότι το θέμα της αναγνώρισης είναι διαφορετικό. Η αναγνώριση και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και η εκπεφρασμένη συνένεση του τρίτου συμβαλωμένου για να ισχύσει. <clears throat> Θέλω λοιπόν να υπάρξει απόλυτη σαφήνεια. Από σήμερα λοιπόν, τι καταλαβαίνω. Για να εφαρμοστεί η απόφαση αυτή, όλα τα προϊόντα από την επικράτεια του Μαρόκου μπορούν να εισαχθούν με βάση τη συμφωνία, ενώ τα γεωργικά προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας δεν μπορούν να εισέλθουν με βάση τη συμφωνία αυτή και θα έπρεπε να υπόκειται σε άλλους δασμούς. Αλλά τι γίνεται τώρα. Οι τελευταίες μας αρχές μπορούν να ξεχωρίσουν το ένα από το άλλο. Γιατί πάνω στο προϊόν, η ντομάτα ας πούμε, λέει προϊόν Μαρόκου. Έχουμε τους κανονισμούς μας που λένε ότι όλα τα νοπά προϊόντα πρέπει να, πρέπει, να, έχουν σήμανση με τη χώρα προέλευσης. Θέτω λοιπόν το ερώτημα, ξέρουμε να τα ξεχωρίσουμε. Άρα θα έπρεπε τώρα, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, να έχουν χωριστή σήμανση τα προϊόντα του, της Δυτικής Σαχάρας. Εγώ αυτά καταλαβαίνω, αλλά πέστε μου κι εσείς για να καταλάβω περισσότερα. Εγώ θεωρώ ότι τα προβλήματα θα είναι ως εξή. Πρώτον, θα έχουμε πολλές αμφιβολίες για τα εισερχόμενα, τα εισαγόμενα προϊόντα. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαφοροποίηση στις ετικέτες, γιατί αλλιώς θα ήταν παράτυπο. Για να το αντιμετωπίσουμε λοιπόν καλύτερα να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας νέας συμφωνίας. Γιατί ναι μεν μπορεί να θεωρείται θεωρητικά εφαρμόσιμη αυτή η συμφωνία, αλλά η πρακτική εφαρμογή της θα είναι πολύ δυσχερής. Επιπλέον, οι σχέσεις μας με το Μαρόκο δεν είναι μόνο εμπορικές, είναι πολιτικές και έχουν μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ισπανία, για την κοινότητα της Ανταλουσίας, από που προέρχομαι. Οπότε λοιπόν εγώ ενώπιον των ε, αβεβαιοτήτων υπό τις, υπό τις οποίες ζουν οι παραγωγοί μας θα πρέπει να διευκρινίσουμε την κατάσταση. Πρέπει να ξέρουμε. Αυτή η ντομάτα που λέει ότι είναι από το Μαρόκο είναι όντως από το Μαρόκο ή μήπως είναι από τη Δυτική Σαχάρα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο. Οπότε να ξαναδώσω το λόγο στους δύο προσκεκλημένους μας για να σχολιάσουν. Ε, διαλέξτε ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος. Δεν μπορώ βέβαια να απαντήσω εγώ στη θέση του συναδέλφου από την εξωτερική υπηρεσία δράσης βέβαια για το τι θα κάνουν, αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο αποφάσεων οδηγεί ουσιαστικά στο ίδιο πρακτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η συμφωνία για τα προϊόντα προέλευση Δυτική Σαχάρα. Η αιτιολόγηση αυτών των αποφάσεων είναι πολύ διαφορετική μεταξύ σα. Καταρχήν, το Γενικό Δικαστήριο είπε πω η Συμφωνία Απελευθέρωση θα μπορούσε να ερμηνευθεί ω εφαρμοστέα και στην περίπτωση τη Δυτική Σαχάρα υπό συγκεκριμένε προποθέσει. Ενώ το ΔΕΚ, υπό το Διεθνέ Δίκαιο, είπε πως δεν μπορεί, το, δεν μπορεί η συμφωνία αυτή να εφαρμοστεί για το λαό της Δυτικής Σαχάρας εκτός αν υπάρχει ρητή συγκατάθεση από πλευράς του λαού αυτού. Άρα λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο είναι διαφορετική και η σημασία των δύο αυτών αποφάσεων ενώ το αποτέλεσμα, το πρακτικό είναι το ίδιο. Κυρία Αγγιλέρα, όντως η απόφαση αυτή έχει να κάνει με τη Συμφωνία Απελευθέρωσης που ενέκρινε το Συμβούλιο το 2012. Γιατί η απόφαση περιορίζεται σε αυτή την προσφυγή που έκανε κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου. Δεν θα επεκταθώ στο καθεστώς ε, ε, που ισχύει μεταξύ και στις διαφορές που έχουμε στα καθεστώτα μεταξύ κάποιων γεωρικών προϊόντων και αλληλευτικών προϊόντων. Ξέρω πως οι συνάδελφοι σήμερα το πρωί σας έδωσαν λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να τονίσω παρόλα αυτά είναι πως οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης ε, δεν οδηγούν σε απαγόρευση ε, εισαγωγών από τη Δυτική Σαχάρα, όχι. Η συνέπεια είναι πως η συγκεκριμένη αυτή συμφωνία απελευθέρωσης που ετέθησε ισχύ το 2012 δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα προέλευσης Δυτικής Σαχάρας. Άρα λοιπόν τα προϊόντα αυτά δεν την χάνουν αυτής της ειδική ε, δασμολογικής αντιμετώπισης που προβλέπεται μέσα στη συνθήκη απελευθέρωσης. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ όλους για τα σχόλια που έκαναν. Να σας ξεκαθαρίσω πως ε, κατανοούμε απολύτως πως πάρα πολλά συμφέροντα πολιτών ε, αυτή τη στιγμή διακυβεύονται. Έχουμε εμπορευόμενους οι οποίοι συνεργάζονται με το Μαρόκο και εμπορεύονται προϊόντα από τη Δυτική Σαχάρα για δεκαετίες για να μην πω περισσότερο και βέβαια διακυβεύεται και η περιουσία τους και θέσεις εργασίας θα χαθούν και όλα αυτά ε, τα κατανοούμε και μας οδηγούν στο να βιαζόμαστε και να αισθανόμαστε μία πίεση για να δώσουμε μία κατάλληλη και νομικά στερη απάντηση στην απόφαση αυτή του δικαστηρίου. Επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικά περίπλοκη η υπόθεση αυτή γιατί έχουμε αυτές τις ε, νομικές επιπτώσεις όχι μόνο σε αυτή τη γεωργική συμφωνία, ε, στη συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα, αλλά και για άλλες δύο αποφάσεις, οι οποίες επαναλαμβάνω ακόμα δεν έχουν εκδικαστεί. Οπότε, σε πολιτικό επίπεδο ε, το θέμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και βέβαια είναι πολύ ευαίσθητο και για τις ίδιες τις αρχές ε, του Μαρόκου και αυτό πρέπει να το λάβουμε δεόντως υπόψη και όπως έχω υπογραμμίσει αρκετές φορές, εμείς δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε, να εμποδίσουμε με οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία του ΟΗΕ επειδή θα επιλέξουμε κάποια συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Αντίθετα, θέλουμε να δούμε πώς γίνεται επιλέγοντας κάποια κατάλληλη αντιμετώπιση να βοηθήσουμε να ξαναρχίσει η ειρηνευτική διαδικασία και ξέρω πως είπα η εκπρόσωπος θα δείξει κάθε ενδιαφέρον έτσι ώστε να αναζωπυρώσει αυτή τη διαδικασία του ΟΗΕ όσο μπορεί. Και νομίζω ότι ίσως έτσι απάντησα και στα σχόλια που έγιναν από τον κύριο Μποβέ. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε στην ειρηνευτική διαδικασία του ΟΕΕ, τη στηρίζουμε, αλλά δεν έχουμε δικό μας ρόλο και καθοδητικό ρόλο και την ευρύτερη κυριαρχία την έχει στο σημείο αυτό ο ΟΗΕ ε, για τις αποφάσεις που θα λάβει. Τώρα, κατά πόσο σκεφτόμαστε μια νέα συμφωνία. Δεν είναι αυτή η λύση που προτιμάμε. Θα προτιμούσαμε μια τροποποίηση της υφιστάμενης συμφωνίας. Για, γεωργική, λοιπόν, για την απελευθέρωση για τα γεωργικά προϊόντα να κάνουμε μια τροποποίηση ε, στείνοντας αυτό που μας ζήτησε το δικαστήριο, δηλαδή κάτι το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, ε, μια σωστή νομική βάση έτσι ώστε οι δασμοί αυτοί να εφαρμόζονται και για την επικράτεια της Δυτικής Σαχάρας με μία διατύπωση η οποία αν θυμόσαστε κι εσείς χρησιμοποιήσαμε και στην περίπτωση της ε, συμφωνίας για τα λευτικά προϊόντα όπου μιλήσαμε για επικράτεια η οποία βρίσκονται υπό μαροκινή διοίκηση το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ε, μιλάει για τη Δυτική Σαχάρα, εδάφη λοιπόν τα οποία διοικεί το Μαρόκο. Αυτό ε, θα πρέπει να το δούμε και με τους Μαροκινούς, να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Βεβαίως, άλλο το τι θα κάνει κανείς νομικά και άλλο το τι θα καταφέρει σε πολιτικό επίπεδο. Θα πρέπει και αυτό να το δούμε. Ε, έχει να κάνει με αυτή την ε, ανάγκη έκφρασης συγκατάθεσης που είναι ένα σημαντικό τμήμα της αιτιολόγησης της απόφασης. Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε μια καλή λύση για το συγκεκριμένο σημείο που δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποια θα είναι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή τη φάση των διερευνητικών επαφών που έχουμε. Τουλάχιστον όχι στις τεχνικές συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αλλά σίγουρα χρειάζεται, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Να σας μιλήσω λίγο και για το χρονοδιάγραμμα. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να δώσω συγκεκριμένες ε, ημερομηνίες, αλλά επειδή γνωρίζουμε ποια είναι η οικονομική κατάσταση και το πόσο απαραίτητη είναι η σαφήνεια εδώ και η βεβαιότητα για τους εμπορευόμενους, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αγγιλέρα, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι. Κάτι πολύ συγκεκριμένο Το θέμα είναι η ρητή συνένεση. Ποιο δίνει τη ρητή συγκατάθεση εκ μέρου τη Δυτική ε, Σαχάρα, ο εκπρόσωπο του Πολυσάριο, γιατί εκεί θα υπάρξει το πραγματικό πρόβλημα στην πραγματικότητα. Να υπάρχει ρητή συγκατάθεση, αλλά πιανού. Ποιο είναι αυτό ο οποίο δίνει ρητή συγκατάθεση εξ ονόματο τη Δυτική Σαχάρα. Και κάτι ακόμα. Πώς μπορεί η Δυτική Σαχάρα αυτή τη στιγμή να μπορεί να εισάγει προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να, προϊα... Ε, να ε, πουλά με διαφορετικό δασμό, όχι με προτιμησιακούς δασμούς σαν αυτούς που έχει το Μαρόκο, αλλά με διαφορετικό δασμό και με σήμανση που θα λέει Δυτική Σαχάρα. Ισχύει αυτό, συμβαίνει, υπάρχει ε, τέτοια δυνατότητα. Διότι εγώ πιστεύω ότι όσο δεν διευκρινίζεται το νομικό καθεστώς, αυτό θα είναι το πρόβλημα. Ότι θα μπορούν να συνεχίσουν να εισάγονται τα προϊόντα, αλλά δεν θα υπάρχει σαφής διαφοροποίηση. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει, αλλά υπάρχει δυνατότητα για επισήμανση Δυτική Σαχάρα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πρόβλημα, αν δεν υπάρξει κάποια νομική λύση. Ε, αλλιώς θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση ε, μέσω της ε, ε, συμφωνίας σύνδεσης στην Αλία, που είναι τελείως διαφορετική. Ο κύριος Μπόβε. Λοιπόν, για να πω κάτι περισσότερο επί του ιδίου μήκου κύματος. Η κύρια είσοδος των Ε, των προϊόντων αυτών ε, κυρίως της ε, τομάτας είναι το Πορβάνδο και η κύρια αγορά είναι το Περπινιό. Υπάρχουν τρεις επιχειρήσεις που κατέχουν το 75% της αγοράς ντομάτας στο Μαρόκο και οι οποίες τις εξάγουν. Και το 75% των εξαγωγών του των εξαγωγών της Δυτικής Σαχάρας είναι ε, ε, το κατέχουν τρεις εταιρείε. Η Deal και Azura που είναι γαλλικές και άλλη μία. Οι εταιρείε αυτές, η Deal και Azura, παράγουν ε, τα φρούτα αυτά, παράγουν αυτά τα νοπά προϊόντα στη Δυτική Σαχάρα. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Μία επιχείρηση που την ξέρουμε και που παράγει και από τις δύο πλευρές, και στην Ισπανία και στη Δυτική Σαχάρα, στην Ισπανία λέει ο δεν έχουμε καμία δυνατότητα να ξεχωρίσουμε διότι αν εξάγουμε το δικό τους όνομα δεν θα μας πούν ε, από πού προέρχονται τα προϊόντα. Υπάρχει ένα πρόβλημα νομικό. Εάν εισάγονται προϊόντα, μπορούμε να τις εντοπίσουμε και να πούμε ότι είναι κατά παράβαση της απόφασης του δικαστηρίου. Γιατί μπορεί να γίνει απάτη, δηλαδή να πούνε ότι είναι από την ε, επικράτεια του Μαρόκου θα πρέπει να υπάρξουν κάποια προσωρινά μέτρα μέχρι να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται σωστά αυτός ο διαχωρισμός. Θα πρέπει δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτές να δεσμευτούν και είπαμε ότι είναι δύο ή μάλλον τρεις οι κυριότερες, τις ξέρουμε, οι εταιρείε αυτές πρέπει να υποστούν την ε, πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επιβάλλουν να δηλώνουν από πού προέρχονται τα προϊόντα τους. Αυτό είναι προϋπόθεση για μια μεταγενέστερη λύση. Σαδωρά. Θέλω να επιμείνω γιατί νομίζω ότι δεν μου απαντήσατε στην ερώτηση, τις ερωτήσεις που σας έκανα και η πρώτη ερώτηση ήταν πώς θα σεβαστείτε τις αποφάσεις ε, των κατοίκων της Δυτικής Σαχάρας και τι σκοπεύετε να κάνετε και το κατά πόσον τηρείται η απόφαση. Δηλαδή, αν το Μαρόκο σταμάτησε να διαθέτει στην κινητική αγορά προϊόντα τα οποία παράγονται στη Δυτική Σαχάρα σαν να είναι προϊόντα Μαρόκου. Και πώς ελέγχεται η εφαρμογή της απόφασης, τι έλεγχοι υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω και πάλι το λόγο στους προσκεκλημένους μας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το ρόλο των πολυσάριων, η απόφαση του δικαστηρίου δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτό η απόφαση του δικαστηρίου λέει ότι πρέπει να έχουμε τη συγκατάθεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας και από εκεί και πέρα τίποτα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να κάνουμε και κάτι σε εσωτερικό επίπεδο και σε διαβούλευση με τους εταίρους μας για να δούμε πώς μπορούμε να σκεφτούμε το θέμα αυτό. Δεν έχουμε καταλήξει κανένα συμπέρασμα, δεν έχουμε καν ξεκινήσει συζήτηση. Θα πρέπει να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά τις τεχνικές πτυχές, για το τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, καταρχάς να σας ε, υπενθυμίσω ότι αυτό που θέλουμε είναι μια βιώσιμη λύση μακροπρόθεσμα. Και βιώσιμη λύση η οποία στόχο θα έχει η νομική βάση να είναι για την εφαρμογή των προτιμησιακών ε, ε, δασμών. Ε, δεν υπάρχει τέτοια νομική βάση αυτή τη στιγμή για τα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας. Το δικαστήριο είπε ότι αν θέλετε να έχετε προτιμησιακό καθεστώς, τότε αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνετε και υπάρχουν μία σειρά από κριτήρια και θέματα τα οποία θα πρέπει να πληρούνται, κυρίως το θέμα της εγκατάθεσης. Και αυτό λοιπόν είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει μακροπρόθεσμα. Και γι' αυτό έγιναν και κάποιες τεχνικές συζητήσεις. Εν τω μεταξύ βεβαίως πρέπει να επιληθεί ε, και το ζήτημα να δούμε ποιες είναι οι καλύτεροι πίστη προσδοκίες των εμπόρων, ε, των ε, συμβάσεων που υπεγράφησαν καλή την πίστη, ε, δεδομένη της κατάστασης που είχαμε στο παρελθόν. Είναι λεπτό το ζήτημα και το γνωρίζουμε. Και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ και πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι θέλουμε να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο στις σχέσεις μας με τους εταίρους μας από πλευράς Μαρόκου. Και να αποφύγουμε να υπάρχουν οποιασδήποτε διαταραχές, οποιασδήποτε μορφής στις σχέσεις μας. Υπάρχουν συνέπειες, το ξέρουμε. Υπάρχουν συνέπειες της απόφασης στις οικονομικές ε, συναλλαγές και φυσικά αυτό δεν ε, εξυπηρετεί κανέναν. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία τώρα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω τώρα. Ε, διότι δεν έχουμε καταλήξει σε συμπεράσματα, αλλά και γιατί νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απαντά και ε, επ' αυτών και όχι η Υπηρεσία εξωτερική Δράσης. Υπάρχουν μία σειρά από ε, στοιχεία τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε ώστε να είναι πρακτικά όλα αυτά και η βάση και της απόφασης. dziękuję. W Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι με το σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος συζήτησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μια φορά ακόμα τους προσκεκλημένους μας. Θα ήθελα να σας πω που σας ευχαριστώ και για τις παρουσιάσεις που κάνατε και για τις γνώμες που ακούστηκαν εδώ και το θέμα αυτό παραμένει ανοιχτό. Θα επανέλθουμε και θα το συζητήσουμε και σε μεγαλύτερο βάθος. Να σας πω τώρα λοιπόν πώς μπορούμε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης να το κλείσουμε και Πάλι σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ήταν πραγματικά πολύ ζωντανή. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε για τα αντίμετρα που ενδεχομένως θα λάβουν οι ΙΠΑ μετά την απαγόρευση που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο βόλιο που έχει υποστεί ορμονοθεραπεία. Στις 20 Δεκεμβρίου το Προεδρείο της ε, Υπουργείου Εμπορίας της, ε, η, με συγχωρείτε, η πολιτική ηγεσία του πολιτικού του του Υπουργείου Εμπορίου της Ευρωπαϊκής της, τον ΗΠΑ μίλησα για μια σειρά από αντίπεινα που θα λάβουν οι ίπα για τα μέτρα παγόρευσης για τις ε, εισαγωγές ε, αμερικανικών προϊόντων ε, βόλου. 20 Δεκεμβρίου λοιπόν 2016 είναι η ημερομηνία στην οποία ήδη αναφέρθηκα και πρέπει να σας πω πως η απόφαση αυτή ε, ελήφθη ε, μετά από προσφυγή εκπροσώπων του Βόλου Κλάδου στις Ηνωμένε Πολιτείες, όπου ε, θεωρούν ότι περιορίζεται η πρόσβαση των Αμερικανών στην αγορά βοήου και πρέπει να σας πω ότι η κοινοποίηση αυτή από το γραφείο του εμπορικού εκπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε για ε, εμπορικές κυρώσεις που μπορεί να φτάσουν σε ύψος τα 116,8 εκατομμύρια ε, δολάρια το χρόνο. Το τελευταίο μέτρο της ε, διαδικασίας θα λήξης της 22 Φεβρουαρίου, δηλαδή της δημόσιας διαβούλευσης του 2017 και μετά το γραφείο αυτό είναι στη διακριτική του ευχαίρεια να λάβει μια απόφαση σχετικά με τη δράση που θα αναλυφθεί ακολουθώντας τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης. Μετά από αίτημα των ε, σοσιαλιστών ε, οι συντονιστές στην Επιτροπή Γεωργίας αποφάσισαν πως δεδομένες αυτής της ε, απειλής για νέες κυρώσεις από τις Ευρωπαϊκές ε, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες πως θα ήθελαν να μας κάνετε μια παρουσίαση για το κατά πόσο αυτά τα αντίμετρα είναι πιθανόν να επιβληθούν ή όχι, τι φύση, ποια θα είναι η φύση τους και πώς αυτό θα επηρεάσει με τη σειρά του τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα η DG Agri έχει ήδη καταθέσει ένα έγγραφο το οποίο ε, συμπεριλαμβάνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και έχει κυκλοφορήσει αυτό σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας σήμερα. Έχουμε τον κύριο Τζον Κλάρκ που είναι διευθυντής στην Γενική Διεύθυνση Agri, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες ε, διευκρινήσεις. Κύριε Κλάρκ, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και θα σας δώσουμε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την κατάσταση, να ξέρουμε κι εμείς πώς έχει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από την συζήτηση που έγινε για το Μαρόκο, νομίζω ότι αυτό το σημείο θα είναι απλό και σύντομο. Είμαι εδώ με τον προστάμενο της μονάδας ε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κύριο Μάιας που είναι ο νομικός μας ε, σύμβολο και τη Μις Μπόλο που είναι ε, νομικός από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Δηλαδή περιτριγυρίζουμε από τους δικηγόρους μου. Πάντα καλή ιδέα σε τέτοιου είδους ε, περιπτώσεις. Να σας εξηγήσω καταρχήν ποιο είναι το ιστορικό αυτής της υπόθεσης γιατί σε αυτή την εποχή με, την, ε, μετά αληθινή εποχή, ε, καλό είναι να ξεχωρίζουμε την πραγματικότητα και την απλή προπαγάνδα. Όπως δείτε και εσείς, το 2009 υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ για να λύσουμε αυτή την ε, ε, αντίθεση που χρονίζει με τη συνεχιζόμενη απαγόρευση στη χρήση ορμονών στην εκτροφή βοηού. Το μνημόνιο αυτό περιέγραψε μια ποσόστοση η οποία ήταν 45.000 τόνοι βόλου, ε, που θα πρέπει να είναι βέβαια ελεύθερο ορμονών και πολύ σημαντικό ήταν μια ποσότηση η οποία δεν ήταν αποκλειστικά και μόνο για τις ΙΠΑ, είναι αυτό ε, που ονομάζουμε έργων όμνης, δηλαδή καλύπτει όλους, ε, οποιαδήποτε δηλαδή χώρα η οποία στέλνει βόλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές οι 45.000 τόνοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι ε, ορμονών. Έργων όμνης λοιπόν, επαναλαμβάνω. Βέβαια, έχει μειωθεί το ποσοστό αυτή της ποσόστοση που έχουν οι ΙΠΑ αυτή τη στιγμή διαθέσιμοι. Είχαν ξεκινήσει καλύπτοντα το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά έκτοτε η Ουρουάη, η Αργεντινή, η Αυστραλία έχουν αρχίσει να κάνουν χρήση αυτή της ποσόστοση, γιατί είναι ανταγωνιστές. Και αυτή την ποσόστοση, επαναλαμβάνω, σήμερα οι Αμερικανοί καλύπτουν μόνο κατά το 1 τρίτο Άρα λοιπόν ο κλάδος του βοήου στις ΕΠΑ ε, δυσαρεστήθηκε με αποτέλεσμα πέρσι το φθινόπωρο να προσφύγουν στο γραφείο αυτό ε, ζητώντας μια αναθεώρηση της ποσόστοσης και ζήτησαν μια επανεισαγωγή κάποιων εμπορικών κυρώσεων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης ζήτησαν και την ε, κατάργηση του μνημονίου. Μη αναφερθήκατε εσείς σε μια διαδικασία που έλαβε χώρα πρόσφατα στην Ουάσιγκτον, όπου έγινε μια δημόσια ακρόαση στις 15 και 16 Φεβρουαρίου. Εκεί κλήθησαν οι εμπλεκόμενοι για να σχολιάσουν ποια προϊόντα ενδεχομένω θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε ένα κατάλογο κυρώσεων που θα ε, λάβουν οι ΙΠΑ ε, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω τώρα μέχρι τις 2 Μαρτίου είχαν χρόνο για σχόλια ε, επιχειρήματα, αποδοχή ή απόρριψη αυτών. Τώρα θα πρέπει η Αμερικανική Διοίκηση καταρχήν να αποφασίσει αν θα διατηρήσει την ποσόσταση και το μνημόνιο ή αν θα τα απαρνηθεί προχωρώντας μετά στην εισαγωγή εμπορικών κυρώσεων ύψους 116 εκατομμυρίων δολαρίων κατ' Επαναλαμβάνω κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση ούτε από την προηγούμενη Αμερικανική διοίκηση, ούτε από τη νέα η οποία ακόμα δεν έχει ε, τοποθετηθεί πλήρους. Ξέρετε πως η Αμερικανική κυβέρνηση, δηλαδή το γραφείο αυτό, έχει την απόλυτη διακριτική ευχαίρεια να αποφασίσει εάν θα αποσυρθεί από το μνημόνιο και εάν αφόσον το αποφασίσει πότε. Οπότε επαναλαμβάνω πως απόφαση δεν έχουν λάβει και δεν αναμένεται απόφαση ε, μέχρι τουλάχιστον να τοποθετηθεί νέος Υπουργός Εμπορίου ΣΥΠΑ. Εμείς παραμένουμε σε επαφή με την Αμερικανική διοίκηση, θα το κάνουμε και τις επόμενες εβδομάδες και πάντοτε η θέση μας ήταν πως είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε οποιαδήποτε ανησυχία διακατέχει την Αμερικανική κυβέρνηση για το πώς λειτουργεί ε, αυτό το μνημόνιο για το βόιο το οποίο δεν έχει υποστεί ορμονοθεραπεία και πάντοτε, και το υπογραμμίζω αυτό, Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Πάντοτε έχουμε συμμορφωθεί απόλυτα και με το πνεύμα και με το γράμμα του, νο... του μνημονίου που είναι ουσιαστικά μια συμφωνία μεταξύ ΕΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εμείς με κάθε πτυχή αυτού του μνημονίου πάντα έχουμε συμμορφωθεί ε, αντίθετα με τα επιχειρήματα που έχει εκφράσει ο κλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επίσης και κάποια μεμονωμένα άτομα της Αμερικανικής Διοίκησης. Εάν, εάν αποφασίσουν η να αποσυρθούν από τη συμφωνία αυτή, που επαναλαμβάνω ε, έχει απόλυτο δικαίωμα να αποφασίσει, τότε αυτό θα εκινήσει μία περίοδο χάριτος εξι μηνών, κατά την οποία η ποσόστοση και το εμπόριο παραμένουν ως έχουν, και κατά την οποία δεν μπορεί να επιβάλλει εμπορικές κυρώσεις η αμερικανική πλευρά και μόνο μετά από έξι μήνες μπορεί να επιβάλλει κάποιες κυρώσεις. Εμείς θεωρούμε πως οι Αμερικάνοι θα σεβαστούν αυτές τις διεθνείς ε, υποχρεώσεις που έχουν και θα σεβαστούν την εξάμεινη αυτή προθεσμία. Εάν βεβαίω οι ΙΠΑ αποφασίζουν να αποσυρθούν από το μνημόνιο χωρίς να έχουμε φταίξει εμείς και να εισάγουν ε, να επιβάλλουν κυρώσει θα το θεωρούσα αρνητικό βήμα στι εμπορικέ σχέσει που έχουμε, αλλά δεν φτάσει και το τέλο του κόσμου. Αλλά σίγουρα δεν είναι ένα βήμα το οποίο μπορεί να μας χαροποιήσει. Νομίζω πως σήμερα είναι αρκετά πρόημο να ε, προσπαθήσουμε να προκαταβάλουμε την θέση την οποία θα λάβει η νέα Αμερικανική διοίκηση και νομίζω ότι αντίστοιχα δεν μπορώ να σας δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες σήμερα για το τι θα κάνει ενδεχομένω ή όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μη γνωρίζοντας ποια θα είναι τα, ποιες θα είναι οι αποφάσεις της νέας ε, κυβέρνησης. Αυτό που μπορώ να κάνω, να σας υποσχεθώ πως θα είστε πάντα ενήμεροι σε κάθε φάση αυτής της διαδικασίας για το θέμα. Και με μεγάλη χαρά θα επιστρέψω εδώ για να τα ξαναπούμε. Εάν έχουμε οποιασδήποτε εξελίξεις. Δευτερόφυγη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Έχουμε λοιπόν κάποιους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Μποβέ καταρχάς. Χαίρομαι με την συνόψηση που είναι πολύ σωστή από πλευράς της Επιτροπής και δεν ενδέχεται, δεν ε, μπορεί να προκαλέσει παρερμηνίες. Αλλά μου προκαλεί και κάποιες σκέψεις. Η πρώτη είναι ότι δεν πρέπει να επανέλθουμε στο 2009 αλλά στο 1997 και σε αυτό το πάνελ στον ε, ΠΟΕ που οδήγησε καταδίκη της Ένωσης το 1998 λόγω άρνησης εισαγωγής βοήου με ορμόνες και μετά από 12 χρόνια υπερβολικής ε, φορολόγησης 70 ε, ευρωπαϊκών προϊόντων θυμάμαι ότι επιτέλους ε, εγκρίναμε αυτή τη συμφωνία γιατί ήταν τελικά το κλείσιμο των διαφωνιών. Όμως, τι διαπιστώνουμε τώρα, δεν αξιοποίησαν αυτή την ποσόστοση πήραν άλλοι ένα μεγάλο τμήμα της ποσόστοσης και θέλουν να διπλασιάσουν τώρα αυτήν την, ε, αυτήν την ε, ποσόστοση. Δηλαδή θα είχαμε τι τύπ στο τομέα των, ε, του βοήου. Αν προσθέσουμε και άλλες 45.000 τόνους, συν τις 50.000 που δόθηκαν μέσω του ΣΕΤΑ και ότι θα διαπραγματευτούμε με το Μερκοσούρ, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να εκτρέφουμε βοηδή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μπορούμε να κλείσουμε το μαγαζί. Δεύτερον, κάτι που είναι πολύ σημαντικό επί της ουσίας, πέρα από την αγορά βοήου, υπάρχει ένα πρόβλημα ουσίας που δεν θα επιληθεί όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιδείξει πιο επιθετική στάση έναντι των διεθνών κανόνων του ΠΟΕ για την αντιστροφή ε, του άχθους της απόδειξης. Τι εννοώ. Όποιος βάζει ορμόνες στο βόλιο δεν έχει αυτό την ευθύνη να αποδείξει ότι δεν είναι επικίνδυνο. Πρέπει η άλλη πλευρά να αποδείξει ότι είναι επικίνδυνο. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Εμείς δεν θέλουμε κρέας με ορμόνες. Γιατί οι αρχές μας, οι, επιστημον, οι επιστήμονές μας λένε ότι είναι επικίνδυνο. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι είναι επικίνδυνο. Ενώ οι ΗΠΑ και ο Καναδάς που βάζουν ορμόνες δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα. Έχει αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και αυτός ο κανόνας του ΠΟΕ. Γιατί στα πλαίσια του κόντεξ αλιμεντάριους επιτρέπονται για την εκτροφή, για την κτηνοτροφία οι ορμόνες. Ποιος μας λέει λοιπόν θα σταματήσει έτσι η κατάσταση. Γιατί είναι όλο και χειρότερη. Σήμερα επειδή λοιπόν δεν μπορούν να μας πουλήσουν αρκετό βόλιο, λένε «Ε, θα επιτεθούμε. Ποιο μπορεί να μα πει τι θα κάνουν αύριο. Δεν έχουν κανένα λόγο να σταματήσουν. Το πρόβλημα είναι ότι υπογράψαμε μια συμφωνία με ένα συγκεκριμένο τμήμα κρέατο χωρίς ορμόνες για να σταματήσει αυτή η διαμάχη. Αλλά μονόπλευρα οι ΗΠΑ όποτε θέλουν το ξανανοίγουν το θέμα. Πρέπει να σταματήσει κάποτε αυτό. Πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί του διεθνού εμπορίου που να εμποδίζουν αυτό το διαρκή εκβιασμό που επιτρέπει να γίνει αυτό που επιδιώκουν σήμερα οι Ηνωμένε Πολιτείες. Για μένα το θέμα είναι ευρύτερο από το θέμα που συζητάμε σήμερα. Είναι ένα θεμελιώδες θέμα των ε, διεθνών εμπορικών συναλλαγών με τους εταίρους μας, ιδιαίτερα για τα θέματα τροφίμων και ιδιαίτερα για το βόλιο. Κάθε φορά σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες που προτείνονται Έχουμε το θέμα του βοήου. και τις δυσχέρειες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι δικοί μας κτηνοτρόφοι αν γίνουν υπερβολικές εισαγωγές βοήου. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις ορμόνες. Μιλάω γενικότερα για το βόηο. Και αν προσθέσουμε και τις ορμόνες τώρα, το θέμα γίνεται ακόμη πιο οξύ. Φυσικά πρέπει να είμαστε Συνεπεί, Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε. Πρέπει να είμαστε ανυποχώρητοι. Γιατί οι καταναλωτέ μα δεν θέλουν ορμόνε. Υπάρχει το θέμα των δασμών, αλλά υπάρχει το θέμα των κανόνων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στι διεθνεί σχέσει. Υπενθυμίζω έτσι για την ιστορία ότι οι Αμερικανοί με, τις, ε, με τους κανόνες που είχαν για το θόρυβο σκότωσαν το αεροσκάφος Concorde. Δεν είναι βέβαια γεωργικό προϊόν το Concorde, αλλά να θυμηθούμε τι μπορούν να κάνουν. Όπως είπε και ο Ζωζεμποβέ, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, λένε πρώτα η Αμερική τώρα. Θα κάνουν λοιπόν ό,τι μπορούν, τόσο ώστε να είναι πρώτα οι Αμερικάνοι, να μπορούν πρώτα εκείνοι να εξάγουν. Και χωρίς κανένα εμπόδιο. Πρέπει λοιπόν και εμεί να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πρέπει να προστατευθούμε κατά αυτών των χειρισμών που οφείλονται σε αυτό το μυθομανή που έχουν πρόεδρο. Πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε μεγάλη αλληλεγγύη για να καταφέρουμε να επικρατήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική της παρουσίαση, σαφέστατη. Μία σύντομη συγκεκριμένη ερώτηση υπάρχει δυνατότητα μεταξύ, α, για άλλε χώρε αντί των ΗΠΑ να συμπληρώσουν την ποσόσταση όπω μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Αυστραλία για παράδειγμα θα μπορούσε να ε, έχει αντίστοιχη ποσόσταση, αλλά είναι αδύνατο για του δικού μα του εξαγωγείς να εξάγουν στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την Επιτροπή και τον κύριο Κλάρκ τον Διευθυντή για την ανάλυση του προβλήματος. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έγιναν καθαρός εισαγωγέας κρέατος και αυτό φυσικά σημαίνει ότι πιέζονται πολύ και αναζητούν συνεχώς ε, νέους τρόπους ε, διεξόδου στην αγορά. Ε, όπως αναφέρθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω, εμεί πρέπει να σεβαστούμε τη συμφωνία και πρέπει να υπερασπιστούμε και του εαυτού μα. Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι η εξή. Ε, Βλέποντα το εμπορικό ισοζύγιο Ευρώπης-ΗΠΑ, κυρίω ε, στον αγροδιατροφικό τομέα, από πλευρά ε, κινδύνων και πιθανών επιπτώσεων από πλευρά Αμερική για τα ε, προϊόντα μα, τι δυσκολίε αναμένετε να αντιμετωπίσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάουσλινγκ. Για μένα το θέμα που τίθεται δεν μπορούν να παράγουν οι Αμερικάνοι κρέας χωρίς ορμόνες. Είναι αδύνατο δηλαδή. Δεν είναι πια σε θέση. Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν μπορούν να εξαγάγουν στα πλαίσια της ποσόστοσης. Εάν τα προϊόντα τους δεν είναι πια ανταγωνιστικά, και το μόνο που έχουν να λένε είναι πρώτα η Αμερική και θα ξεκινήσω εμπορικούς πολέμους, εντάξει τότε. Αλλά και υπό την ε, κυβέρνηση Ομπάμα είχε, είχαν ήδη να ξεκινήσουν τα προβλήματα. Είχαν, ήδη ξεκινήσει τα προβλήματα. Τώρα όμως είναι ακόμη χειρότερη κατάσταση. Έχουμε κάνει καθόλου συζητήσεις με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση. Και ποια είναι η στάση τους. Δηλαδή είναι σοβαρή αυτή η απειλή. Η είναι, η... πρόκειται να εφαρμοστεί ή είναι απλώς έτσι κομπασμοί. Και με τι μας απειλούν. Μας απειλούν με αντίπεινα σε γεωργικά προϊόντα. Ή μήπως και για μοτοσικλέτες ας πούμε. Δηλαδή έχουν σοβαρά την πρόθεση να ξεκινήσουν εμπορικό πόλεμο. Ή απλώς θέλουν να τροποποιηθεί η ποσόστοση του βοήου. Καλά, φυσικά βέβαια ε, ω χειρονομία δεν μπορεί παρά να μας δυσαρεστεί. Μαγκίνες, η Αντιπρόεδρος κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Κλάρκ ε, που μας ε, ανέλησε την υπόθεση και τον τρόπο με τον οποίο μας παρουσίασε τα στοιχεία. Ε, θα μπορούσε να είναι πολύ ανησυχητική η εξήγηση και δεν αφορά μόνο το βόλιο κρέο. Τα προϊόντα τα, στα οποία θα μπορούσε να επιβάλλει ίσως πολύ ψηλούς δασμούς ε, η Αμερική θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Ε, υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος προϊόντων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από αυτή την επιβολή δασμών και η καθαρή παραγωγή στι ΗΠΑ θέλουν να λάβουν δράση. Θυμάμαι τότε που ήταν επίτροπος ο Πίτερ Μάντελσον και ζήτησε να υπάρξει μια συμφωνία παγκοσμίου εμπορίου και ίσως αυτά τα προβλήματα δεν θα είχαν λόγο ύπαρξη αν υπήρχε ε, παγκόσμια συμφωνία. Αυτά βέβαια είναι ιστορίες του παρελθόντος, ε, αλλά θα θέλαμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τις πιθανές συνέπειες για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ακολουθήσουν αυτή την άγουσα. Ε, ξέρουμε ότι ουσιαστικά μιλάμε χωρίς να γνωρίζουμε ε, τίποτα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει, αλλά σίγουρα δεν είναι καλό σημάδι αυτό και δεδομένης και της νέας ε, ε, ε ιστορίας που έχει ξεκινήσει η νέα Αμερικανική κυβέρνηση για την Αμερική που θα έρχεται πάντα πρώτη, σίγουρα θα επηρεάσει τις εξαγωγές και δεν θα το θέλαμε αυτό σε καμία περίπτωση και θα είναι εις βάρος και αυτών που προσπαθούν να κάνουν κάποιο άνοιγμα στην αγορά εκεί. Δεν θα ήθελα να κάνω προβλέψεις και φαντάζομαι ότι ούτε και εσείς θα κάνετε, αλλά θα ήθελα να ξέρω τι αποτέλεσμα μπορεί να έχουμε μετά από αυτό το εξάμεινο και τι συζητήσεις έχετε με την αμερικανική πλευρά. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις για το τι θα μπορούσε ίσως να συμβεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάναγκαν, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θέσω αυτή την ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη θέτω αρκετές φορές. Υποτίθεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να εφαρμόσουμε πολιτικές για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς η εξαγωγή δεκάδων χιλιάδων τόνων βοήου κρέατος συνάδει με αυτό. Δεν λέω αν είναι λάθος ή σωστό, απλώς λέτε ότι σκοπεύετε να κάνετε κάτι για την αλλαγή του κλίματος. Πώς λοιπόν μπορείτε να τα συντεριάξετε αυτά. Και επίσης, ε, μου προξένησε το ενδιαφέρον ο τρόπος που το παρουσιάσατε το θέμα. Αναφερθήκατε στην ε, εποχή μετά από όλη αυτή την ιστορία. Πολλά ψεύδι υπάρχουν στα μέσα ενημέρωση, τα οποία διασπείρουν αρκετοί. Η ιδέα ότι είναι κάτι καινούριο αυτό είναι ε, πραγματικά ιδίε. Ε, ε, ξεκινήσαμε ποτέ από μια εποχή που ο κόσμο έλεγε την αλήθεια. Κοιτάξτε την ιστορία. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η εποχή της αλήθεια και αυτή μπορεί να είναι η εποχή μετά την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύουν αυτά τα πράγματα. Äh, ναι. Το θέμα αυτό βεβαίως ε, αφορά το θέμα του κρέατος με ορμόνες. Αλλά είναι οπωσδήποτε μια ευκαιρία για να θέσουμε τις κόκκινες γραμμές μας που αφορούν την μη αποδοχή του κρέατος με ορμόνες και το, την μη αποδοχή των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε πώς είναι δυνατόν να αμφισβητούν τα δικά μας κριτήρια, τις δικές μας προδιαγραφές. Πώς είναι δυνατόν ορισμένοι να μας ε, αμφισβητούν αυτό το δικαίωμα. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουμε την αποφασιστικότητα, να υπερασπιστούμε την ε, εκπεφρασμένη βούληση των λαών μας ότι δεν θέλουμε ούτε ορμόνες, ούτε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και νομίζω ότι προσπαθούν έτσι κομμάτι το κομμάτι να υπονομεύσουν ε, αυτή μας την εκπεφρασμένη βούληση. Θέλουν, για παράδειγμα, τώρα να αμφισβητήσουν, αμφισβητήσουν το ένα, μετά θα αμφισβητήσουν το άλλο. Θα πρέπει να επιδείξουμε συνέπεια, αποφασιστικότητα είναι ο δικός μας κόσμος, οι δικές μας χώρες, ο δικός μας κόσμος εδώ στην Ευρώπη. Εμείς θα ε, αποφασίσουμε τι επιτρέπουμε να μπει στην αγορά μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να το απονομεύσει. Ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσω τώρα από τον κύριο Διευθυντή να αντιδράσει στις ερωτήσεις και τα σχόλια που μόλις ακούσαμε. Ευχαριστώ. Σημείωσα 9-10 ερωτήσει από διάφορους ε, ευρωβουλευτές. Θα επιχειρήσω να απαντήσω. Το πρώτο βασικό είναι ότι το θέμα δεν είναι βόλιο με ή χωρί ορμόνες. Υπάρχει ενωσιακή απαγόρευση βοήου με ορμόνες. Ισχύει και θα συνεχίσει να ισχύει. Δεν αμφισβητείται. Καθόλου. Να είναι αυτό απολύτως σαφές. Δεύτερον, η στάση της Αμερικανικής κυβέρνησης δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, άρα δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Είναι σε μεταβατική φάση. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η άποψη των αρμοδίων φορέων. Ελπίζουμε να είναι λογική η στάση τους. Ελπίζουμε να αναγνωρίσουν δημόσια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις της ε, στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεννόησης. Γι' αυτό αναφέρθηκα σε στοιχεία και ψεύτικα στοιχεία, γιατί υπάρχουν ε, κάποιες ε, δηλώσεις καθαρά προπαγανδιστικού χαρακτήρα ότι δεν έχουμε τηρήσει τις υποχρεώσεις μας. Θα οδηγήσει σε εμπορικό πόλεμο, όχι δεν νομίζω, μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες ε, δυσάρεστες αψημαχίες αλλά δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να ξεκινήσει νέα διαμάχη, νέες δυσχέρειες τόσο νωρίς μετά την ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ. Αυτά που είπε ο κύριος Μποβέ για την προϊστορία του θέματος ε, έχει δίκιο δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες του ΠΟΕ για το βάρος της απόδειξης. Πρέπει να ζήσουμε με την εφαρμογή τους. Θα θυμάστε, γιατί τότε ήσασταν ακριβώς, ε, θυμόμασταν, ότι ήμασταν στα, ήσασταν εσείς στα χαρακόμματα, αλλά χάσαμε την υπόθεση του ΠΟΕ. Η απαγόρευση των ορμονών στο Βόλιο θεωρήθηκε ότι ήταν ανεπαρκώς επιστημονικά στοιχειοθετημένη. Χάσαμε και πρέπει να υποστούμε τις συνέπειες. Κάποια άλλα θέματα. Ο κύριος Μπόβε είπε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν και την πίτα ολόκληρη και τον ε, σκυλοχορτάτο. Θέλαν κάποιες παραχωρήσεις μέσω του TTIP και κάποιες παραχωρήσεις μέσω του μνημονίου. Όχι. Δεν προτιθέμεθα να αυξήσουμε τον όγκο που επιτρέπεται μέσω του μνημονίου, τον όγκο ΣΑΟΟΝ, θα προτιμούσαμε η μακροπρόθεσμη λύση να προκύψει μέσω του TTIP. Αλλά τώρα το TTIP ε, προφανώς ε, έχει μπει στην κατάψυξη, δεν θα μας δώσει λύση στο εγγύς μέλλον. Κάποιος ρώτησε, νομίζω ότι υπήρξε μια ερώτηση για τις δικές μας εξαγωγές υπόθηκε ότι η Αυστραλία εισάγει μεγάλες ποσότητες και εμείς δεν μπορούμε να εξαγάγουμε στην Αυστραλία. Αυτό ισχύει. Μόνο ένα κράτος μέλος, η Ολλανδία, έχει λάβει την πρώτη έγκριση εξαγωγών στην Αυστραλία που συνεχίζει να εφαρμόζει την ε, απαγόρευση λόγω της ασθένειας των τρελών αγελάδων, της ε, εγκεφαλοπάθειας των βοηδών η Λουθανία, η Ιρλανδία και δύο άλλες χώρες νομίζω έχουν πάρει έγκριση εξαγωγών προς τις ΗΠΑ. Οι άλλοι δεν μπορούν να εξαγάγουν τίποτα. Σωστά το αναφέρετε. Θέλουμε να υπάρχει εμπόριο βοηδών. Οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν αυτήν και άλλες ποσοστώσεις που τους επιτρέπουν να εξάγουν. Εμεί δεν μπορούμε να εξαγάγουμε σχεδόν τίποτα ούτε προς τι ΗΠΑ, ούτε προς την Αυστραλία, ούτε και προς αρκετέ άλλε χώρες. Και τέλο. κάποιες ερωτήσει για τον κίνδυνο κυρώσεων επιπροϊόντων και επιπίων προϊόντων. Κατά τη διαδικασία διαβουλεύσεων, συγγνώμη, δημόσια διαβούλευση που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ νωρίτερα, το 80 μήνα, έδωσαν ένα ενδεικτικό κατάλογο προϊόντων και κλάδων που θα μπορούσαν να υποστούν κυρώσεις. Με βάση προϊόντα επί των οποίων έχουν επιβάλει κυρώσεις και στο παρελθόν. Καλύπτουν τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα, κομμένα λουλούδια, ντομάτες, λουκάνικα, προϊόντα κρέατος, ε, κάποια ζαχαροπλαστικά, μουστάρδες, σούπες, ε, μεταλλικό νερό, συστατικά των κτηνοτροφών, και όπως είπαν και κάποιοι άλλοι ακόμη και τα τσιμπιδάκια για τα μαλλιά και τις μοτοσυκλέτες δεν ξέρω γιατί και επίσης φυσικά το βόιο και το χοιρινό κρέας πολλά προϊόντα λοιπόν από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέλεγαν ορισμένα από αυτά και θα επέβαλαν δασμούς έως και 116 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο σημαντικό ποσό αλλά λάβουμε υπόψη ότι η αξία του βοήου είναι γύρω στο μισό δις. Εν πάση περιπτώσει είναι ενδεικτικός ο κατάλογος που ανέφερα, δεν ξέρουμε. Εάν αποφασίσει να επιβάλλει κυρώσεις η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ποια θα επιλέξει από αυτά τα προϊόντα και ποια όχι. Α, θα ήταν καθαρή μαντία να σας πω ποια από αυτά θα επιλέξουν. Και κάτι τώρα για το εμπόριο βοηθών και την κλιματική αλλαγή. Θα παρακαλούσα τον ε, αξιότιμο Ευρωβουλευτή στη δήλωση του κυρίου Χόγκαν στις δηλώσεις του κυρίου Χόγκαν τις τελευταίες μέρες και χθε που παρουσίασε τα στοιχεία για τον πόρο του 2016 τέθηκε μια ερώτηση γι' αυτό από τον τύπο και είπε ο κύριος Χόγκαν ότι η Ένωση προσπαθεί η παραγωγή βοήου να γίνει όσο γίνεται βιώσιμη και γενικότερα η γεωργική παραγωγή ούτω ώστε να σέβεται τους στόχους της ε, Συμφωνίας COP21 για την κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Μποβέ θέλει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι απαντήσεις σας ήταν πάρα πολύ σαφείς, τέλειες, αλλά έχω δύο στοιχεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Καταρχήν για τις κυρώσεις να σας υπενθυμίσω Αν δούμε τι έγινε το 99, 98-99, είχαμε 100% φορολόγηση σε κάποια α, ευρωπαϊκά προϊόντα, για παράδειγμα στο Ροκφόρ για 12 χρόνια. Θυμόσαστε τι είχε συμβεί. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να στηρίξει τα προϊόντα τα οποία ε, φορολογούνται με πλέον 100% φόρο, γιατί δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο ο ΠΟΕ. Θεωρείται δηλαδή εμπόδιο στις το οποίο δημιουργεί μια μη βιώσιμη κατάσταση για όσους είναι τα θύματα αυτών των κυρώσεων. Και για το μηχανισμό που θα στήσετε, θα ήθελα να μου πείτε τι θα συμβεί. Γιατί είναι οι άλλες χώρες οι οποίες μπήκαν ε, σε αυτή την ποσόστοση που δώσαμε. Δηλαδή, τι κάνουνε. Χρησιμοποίησαν τους κανόνες του ΠΟΕ Και είπαν, αφού έχουν δικαίωμα οι ΙΠΑ, γιατί είναι το κράτος που στηρίζεται περισσότερο, ανοίξτε την ποσόστοση και για μας. Και αυτή ήταν η παγίδα. Γιατί πιστεύω πως τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να προστατευτούμε από κάτι τέτοιο. Διαφορετικά μιλάμε για το απόλυτο άνοιγμα. Ένας ένας να μας επιτεθεί με τον τρόπο αυτό, όλοι οι υπόλοιποι ε, το χρησιμοποιούν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να περιορίσουμε το άνοιγμα αυτής της αγοράς, μια και αυτή η ποσόστοση είναι ανοιχτή για όλους. Αν παραμείνουμε ε, σε αυτόν τον ε, κανόνα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αντισταθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαθήκαμε. Άρα λοιπόν το πλέον ευνοούμενο κράτος και ο κανόνας είναι μια παγίδα στην οποία δεν θα πρέπει να πέσουμε, γιατί στην περίπτωση επίλυσης διαφορών δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να χρησιμοποιείται. Διαφορετικά, τι γίνεται. Έχουμε πρόβλημα με τη ΣΥΠΑ και τελικά οι υπόλοιποι ε, βρίσκουν ένα παραθυράκι και μπαίνουν και αυτοί. Και δημιουργεί αυτό ε, προβλήματα, ενώ η αρχική υπόθεση είχε να κάνει μόνο με τις υπόποτε Οπότε καταλήγουμε σε μια πάρα πολύ στρεβλή κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Όπως είπα, δεν έχουμε καμία πρόθεση να διευρύνουμε ε, αυτή την ε, ποσόστοση. Θα παραμείνουν 45.000 ε, τόνους. Φαντάζομαι αυτό σας χαροποιεί. Δεν θεωρώ πως η αρχή του πλέον ευνόμενου κράτους είναι ποτέ παγίδα ή μειονέκτημα εμπορικό. Είναι ένα θεμελιώδες κομμάτι του διεθνούς εμπορικού συστήματος και δεν πρέπει να το αμφισβητήσουμε ή να το αλλάξουμε είμαστε υποχρεμένοι, παρόλο που είναι αυτόνομη ποσόστοση, να την βασίσουμε στη ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους και η πραγματικότητα είναι πως και άλλες χώρες έχουν γίνει συν χρόνο πιο ανταγωνιστικές στην παραγωγή βοηού ελεύθερο από ορμόνες. Για παράδειγμα, γι' αυτό οι Ουρουάκοι και οι Αργεντινοί έχουν κομμάτι αυτής της ποσότητας και αυτό φαίνεται. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να θέσουμε υπό αμφισβήτηση την αρχή του πλέον ευνοούμενου κράτους γιατί μας προστατεύει όλους και τους πιο μικρούς και τους πιο μεγάλους. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως είπαμε ό,τι είχε να υποθεί. Καταφέραμε να παρατείνουμε και τη συζήτησή μας γιατί όπως σας είπα στην αρχή δεν θα γίνει σήμερα ανταλλαγή απόψεων με τους επιτρόπους. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιο συγκεκριμένα τον κύριο Κλάρκ. Βλέπω πως ο κύριος Μποβέ και ο κύριος Κλάρκ αυτή τη στιγμή συνεχίζουν την ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα τώρα να εγκρίνουμε τις συστάσεις ε, τις οποίες ενέκριναν σήμερα οι συντονιστές. Έχετε λάβει το σχετικό κείμενο, γραπτά, και βέβαια το έχετε και σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου. Αν δεν έχουμε αντιρρήσεις, μπορώ να θεωρήσω πως εγκρίθηκαν. Θα τα ξαναπούμε στο Στρασβούργο τη Δευτέρα. Επτά με δέκα και μισή νομίζω ε, μας έχουν προγραμματίσει. Είναι βαρύ το πρόγραμμα. Θα τα ξαναπούμε εκεί. Νομίζω πως η μερίσια διάταξη δεν έχει άλλα σημεία. Καλό απόγευμα και τα ξαναλέμε 13 Μαρτίου και μετά πάλι 21 και 22. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.